Thank you, colleagues. Freedom of press and media. Ελευθερία των μέσων, το τύπου και των μέσων ενημέρωση ανά τον κόσμο. Συγγέντρια κυρία Σάκη. So we start the afternoon with the first consideration. Λοιπόν, είναι η πρώτη εξέταση του σχεδίου έκθεσης για την ελευθερία τύπου και μέσων ενημέρωσης στον κόσμο. Το σχέδιο έκθεσης αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Μόλις όμως είναι έτοιμες όλες οι μεταφράσεις όλες τις γλώσσες, θα τις λάβετε ηλεκτρονικά από τη γραμματεία. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η, τελική, η καταληκτική ε, υποβολής τροπολογιών είναι Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Δίνω κατευθείαν το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τους συναδέλφους και όλους τους εμπλεκόμενους και όλα τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών που συμμετείχαν με ιδέες και προτάσεις στο πρώτο αυτό σχέδιο. Ξεκινήσαμε με ένα έγγραφο συζήτησης. Η διαδικασία ήταν όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο κάνουμε εδώ να είναι καλό αποδεκτό και να είναι εποφελές κυρίως αυτούς που δουλεύουν στα διάφορα πεδία και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Μια σημείωση πριν αρχίσω να κάνω τη σύντομη ε, περίληψη του σχεδίου ε, επέλεξα εσκεμένα το θέμα της ελευθερίας του τύπου και των ε, μέσων ενημέρωσης για το τι θα πρέπει να κάνουμε με βάση μια θεματική ανάλυση. Ε, συγκεκριμένα επέλεξα να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένες χώρες, κυρίως γιατί είναι αδύνατο να τις αναφέρουμε όλες και δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε το πολύτιμο έργο πολλών ε, ομάδων της κοινωνίας των πολιτών που κάθε χρόνο κάνουν τέτοιους καταλόγους. Ξεκινά λοιπόν η έκθεση με τις αρχές και το ρόλο του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρει τη σημασία τους για την ελεύθερη έκφραση και για τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τα προγράμματά μας για να προσθέσουμε στη, στο έργο των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων των δημοσιογράφων και βεβαίως αναφέρουμε ότι θα είμαστε αξιόπιστοι μόνο αν και εμείς είμαστε εντάξει. Θέλω να, ε, να αναφέρω και να θυμίσω ότι η έκθεση αυτή αφορά το εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα αναφερθούμε στο τι τυχόν χρειάζεται να βελτιωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε τους διάφορε απειλέ κατά των δημοσιογράφων, που είναι πολυάριθμες, θα πρέπει να πούμε ότι πολλέ από τι απειλέ και του περιορισμού εξακολουθούν να προέρχονται από τι κυβερνήσει. Μερικέ φορέ με νομική πίεση, αλλά και πολλέ φορέ με την κατάχρηση άλλων νόμων που δεν έχουν σχέση με, την, με τον τύπο, αλλά ε, αντιτρομοκρατικού νόμου ή νόμους εθνική ασφάλεια.

που χρησιμοποιούνται προς εκφοβισμό. Ε, ταυτόχρονα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν άλλοι νόμοι που αφορούν τη δυσφήμιση, τη συκοφάντηση ή τη βλασφημία. Χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν την ελευθερία έκφραση των δημοσιογράφων, πράγμα που οδηγεί σε λογοκρισία και αυτολογοκρισία. Ταυτοχρόνως το θέμα της συγκέντρωσης της ε, ε ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης είναι σοβαρό πρόβλημα. Η έκθεση επίση αφορά τις επιπτώσεις τη ψηφιοποίηση, το τοπίο των μέσων Ενημέρωση ενημέρωσης αλλάζει ταχύτατα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και μία από τι άλλε απειλέ είναι ότι πολύ συχνά οι κυβερνήσει πιέζουν για την, ε, ε, για την ιδιωτικοποίηση τη, μέσω του διαδικτύου. Παρά τα ε, η ψηφιοποίηση ε, προσφέρει ευκαιρίες για έκφραση και πρόσβαση στις πληροφορίες και νέους τρόπους έκφρασης της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Όμως, έχει και νέες ε, δυσκολίες, ανάμεσα, όπως ας πούμε την ασαφή γραμμή ανάμεσα στην πληροφορία και τα, τις ειδήσει αν παρακολουθήσουμε τα προγράμματα και τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δούμε ότι υπάρχουν αρκετές πολιτικές και προγράμματα. Υπάρχει όμως περαιτέρω βελτίωση, ε, περιθώριο για βελτίωση και για να εστιαστούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ε, ένα όραμα με πιο ξεκάθαρους συγκριτικούς δείκτες. Παραδείγματο χάρη, η ΕΦΚΟ και η, υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να συνεργάζονται και να συντονίζουν τη δουλειά τους και να κάνουν συνέργειες και προγραμματισμένο έργο. Αυτό θα πρέπει να δημιουργήσει ένα, μια ad hoc ε, επιτόπου ε, δράση σε συνεργασία με επιτόπιες μικρές οργανώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο στην άμεση γειτονιά της και να δουλέψει για το θέμα της ελευθερίας του τύπου και των μέσων ενημέρωσης στο πλαίσιο των χωρών που βρίσκονται υπό στην πορεία της ένταξης και στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Αν δούμε τα χρηματοοικονομικά μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Πρόθεση των Ανθρωπιών Δικαιωμάτων και τα γεωγραφικά μέσα πρέπει να είναι πιο ευέλικτα για να ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών. Και εδώ δίνουμε ε, έμφαση στο να έχουν σχέση με τις τοπικές οργανώσεις και τη δημιουργία δυνατοτήτων. Να μην συνεχίζεται λοιπόν η σχέση εξάρτησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιτόπου. Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι και ο τύπος και τα μέσα ενημέρωση σε τρίτες χώρες είναι ότι αφού έχουν εκφοβιστεί και έχουν περιοριστεί ε, ε, υπάρχει ατιμορρησία και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, την ατιμορρησία αυτή κυρίως προσφέροντας βοήθεια στην διερεύνηση ε, εγκλημάτων κατά των δημοσιογράφων ή προσπαθώντας να δημιουργήσουμε ένα ταμείο νομικής υποστήριξης, υπεράσπισης και να εξασφαλίσουμε ότι οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να έχουν υπεράσπιση και να μην μπορούν να εκφοβίζονται χωρίς τη δυνατότητα να αντιδράσουν ένας άλλος ρόλος που θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν να συμπεριληφθούν στοιχεία στήριξης το τύπου και των μέσων ενημέρωση όταν βοηθούμε ε, τρίτες χώρες με το εκλογικό του σύστημα παραδείγματο χάρη με την ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στους εκλογικούς οργανισμούς και τον τύπο σε τρίτε χώρε για να εξασφαλιστεί η νομιμοποίηση και η διαφάνεια της ε, εκλογικής διαδικασίας και ω εκ τούτου να υπάρχει περισσότερος έλεγχος από τα τοπικά μέσα ενημέρωση. Μια άλλη πρόταση πριν ολοκληρώσω θα ήταν πολύ χρήσιμο αν η υπηρεσία εξωτερικής δράσης χρησιμοποιούσε καλύτερα την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υφιστάμενες σχέσεις με πολυμερή φόρα όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΑΣΕ και σε οπουδήποτε αλλού σε ολόκληρο το χώρο των Ηνωμένων Εθνών. Και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μέσω της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα δημιουργήσουν μια στρατηγική για τον τύπο και τα μέσα ενημέρωση περιλαμβανωμένου και του ψηφιακού στοιχείου που χρειάζεται για να μπορέσει να υπάρχει ένα καλύτερο όραμα εκ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο για την πρόθεση τη ελευθεροτυπία και τη ελευθερία των μέσων ενημέρωση. Κλείνοντα, θέλω να πω ότι ελπίζω ότι οι σκιώδει εισηγητέ συμφωνούν ότι δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε το έργο τη κοινωνία των πολιτών για να παρουσιάσουμε μια σειρά από αξιολογήσει αναχώρα για την ελευθερία του του Είναι πολύ ευπρόσδεκτες βεβαίως οι προσθήκες σας στην θεματική στο θεματικό σχήμα της έκθεσης και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με πνεύμα συνεργασίας όπως και πιστεύω ότι θα συμβεί έχοντας κατά νου ποιοι είναι αυτοί τους οποίους επιδιώκουμε να προστατεύσουμε και θέλουμε να τους βοηθήσουμε να προωθήσουν την ελευθερία της εκφρασής τους μέσω του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουν εγγραφεί τρεις ομιλητές. Κυρία πρώτη. Ευχαριστώ κύριε. Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπε η συγγήτρια και τη συγχαίρω. Έχει κάνει άριστη δουλειά. Ε, θα δούμε στις τροπολογίες μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θα πρότεινα να ακολουθήσουμε τη συμβουλή σας και θα το κάνω εγώ και ως και του ΕΛΚ, να μην μπούμε σε επιμέρους χώρες Έχουμε κάνει εκθέσεις για τις χώρες γειτονίας ή χώρες με τις οποίες έχουμε εσδήποτε σχέσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουμε αιτήσει εκθέσεις και έχουμε εκεί την ευκαιρία, όπως και το πράττουμε άλλωστε, να αναφερόμαστε σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και σε χώρες με ονοματεπώνυμα. Γιατί τώρα αν αρχίσουμε σε μια τόσο γενική έκθεση να κατονομάζουμε χώρες, θα φτάσουμε σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, εξετάζουμε τα θέματα έτσι γενικά, γιατί για πρώτη φορά αναφερόμαστε και στα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα το σκεφτόμουν και ρώτησα και άλλους. Σε μια τέτοια έκθεση για την ελευθεροτυπία πρέπει να αναφέρουμε και αυτά τα μέσα και νομίζω ότι η απάντηση είναι καταφατική. Διότι αλλιώς θα περιέλθουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε πού είναι ε, ε, το όριο. Ποιος είναι δημοσιογράφος και ποιος δεν είναι. Ας πούμε κάποιος έχει ένα ιστολόγιο, ένα blog γράφει, αλλά δεν είναι δημοσιογράφος και μπορούν τα καθεστώτα να τους φέρονται ε, σαν να ε, ή το δημοσιογράφοι, γιατί τους, βρίσκουν, τους θεωρούν πάρα πολύ επικίνδυνους και με εξουσία. Δηλαδή, ε, χρειαζόμαστε συζήτηση, πρέπει να γίνει αυτή, θα δούμε τι θα προκύψει στις επίσημες τροπολογίες. Τώρα είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αλλά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνουμε και αυτά τα μέσα στην έκθεση είναι καλό από μόνο του. Λοιπόν, υποστηρίζω αυτή τη γενική προσέγγιση και τα όσα είπε η συγκήτρια, ότι δεν αναφέρουμε ούτε χώρε ούτε περιπτώσεις, γιατί έχουμε άλλα φόρα για να το κάνουμε αυτό και θα παρακαλούσα να παραμείνει και αυτό το στοιχείο και τα κοινωνικά μίντια λοιπόν και η ψηφιοποίησή τους στην έκθεση. Αυτά προς το παρόν. Και τελείωσα. Thank you. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας. Ο τίτλος, οι υπότιτλοι που έχει συμπεριλάβει η συγγετρία μας δίνουν ένα πολύ καλό πλαίσιο εντός του οποίου μπορούμε να κινηθούμε πολύ σωστά λαμβάνει υπόψη τα θέματα της ψηφιοποίησης και τις διάφορες παραμέτρους τους. Όμως πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τον τίτλο της στρατηγικής και να δούμε ποιες είναι οι στρατηγικές μας απαιτήσεις. Οι αλλαγές στην επικοινωνία πρέπει να αντικατοπτρίζονται και στι απαιτήσει ελευθερία του τύπου και να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια στρατηγική σχετικά. Ο, η εισηγήτρια προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται στενότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να αναφέρεται σε αυτό το σημείο. Ίσως θεωρήθηκε αυτονόητο, αλλά το προφανές καμιά φορά καλό είναι να αναφέρεται. Από τότε που το Ευρωκοινοβούλιο έχει αναλάβει διαφορετικό, σημαντικότερο ρόλο στην σύνταξη εκθέσεων και επηρεάζει ακόμη και τη σύναψη συμφωνιών, οι συμφωνίες αυτές πάντοτε έχουν κριτήρια επιλεξιμότητας, συγκριτικές αξιολόγησης. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και το Ευρωκοινοβούλιο θα να συνεργάζονται και μεταξύ του. Και αυτό πρέπει να τονιστεί επαρκώ. Ούτω ή άλλω, διεθνεί συμφωνίε που να μην συμπεριλαμβάνουν σαφείς μηχανισμούς παρακολούθησης μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, ακόμα και για την επιλεξιμότητα, την αιρεσιμότητα, όταν να μιλάμε για την ε, ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αυτό θα ήταν ε, κάτι που θα το θέλαμε. Στην έκθεση αυτή θα έπρεπε να είμαστε κάπως πιο έντονοι στη διατύπωση. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ρήμα considers. Θεωρεί, ε, ίσως ένας εντονότερος όρος να ήταν προτιμότερος. Είμαστε κάπως χαλαροί εδώ στη διατύπωση. Κάπως επικείς στις συστάσεις μας. Λόγω χάρη για τη χρηματοδότηση, για την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι πολύ καλές οι προτάσεις σας, κυρία Σάκη, στα σημεία αυτά, αλλά σε ό,τι αφορά την πολυφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, Νομίζω ότι αναλύονται τα θέματα αυτά με τρόπο ικανοποιητικό, κυρίως στο έγγραφο εργασίας. Γι' αυτό στον τίτλο, στο υποκεφάλαιο για τη στρατηγική, θα έπρεπε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση ακριβώς τη συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα χέρια λίγων. Βέβαια, πρέπει να πω ότι διαφωνώ και ίσως να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Διαφωνώ με αυτό που είπε η σκιώδης συγκήτρια του ΕΛΚ, ότι δεν υπάρχει λόγος να κατονομάζονται χώρες ή να παρεθνούνται χώρες. Εκεί όπου οι εξελίξει ε, για τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν ήταν θετικέ. Δεν λέω να υπάρχει διεξοδικό κατάλογο, όμω καλό θα ήταν οι χώρε όπου είχαμε δραματική επιδείνωση, δραματική επιδείνωση των συνθήκων για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου υπήρξε υποβάθμιση του ρόλου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι κακό να κατονομαστούν. Συμφωνώ ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προασπίζεται την ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό θα πρέπει να το προωθήσουμε ως ιδέα και ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτουμε εργαλεία και για τα ίδια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά να αξιοποιούνται τον Φεβρουάριο η Επιτροπή για τις Ελευθερίες του Πολίτη ενέκρινε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία για το ίδιο ακριβώς θέμα, δηλαδή την ελευθερία του τύπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση αυτή είχαμε σημαντικά θέματα που θα περάσουν στην Ολομέλεια του Μαΐου. Νομίζω λοιπόν ότι η συμπερίληψη και η μνήα της έκθεσης αυτής στην έκθεση που τώρα εξετάζουμε θα ήταν πολύ θετική κίνηση. Νομίζω πάντως ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας κυρία Σάκη όπως είπα και ελπίζω ότι θα τη δουλέψουμε κι άλλο την έκθεση αυτή. Πάνω απ' όλα ελπίζω να έχουμε περισσότερα χειροπιαστά παραδείγματα και αναφορές των χωρών των σημείων όπου έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώ γύρω στις 5 θα πρέπει να φύγω για να επιστρέψω στη χώρα μου. Δεν θα έχω το χρόνο να ακούσω τις απαντήσεις ε, της εισηγήτριας αλλά ε, ο βοηθός μου θα είναι εδώ για να καταγράψει όλες τις απαντήσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άτκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η ουσία της ε, έκθεσης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Δεν μπόρεσα να την μελετήσω παρά μόνο σήμερα το απόγευμα, αλλά αυτό που μόνο με ανησυχεί είναι υπάρχει ένα στοιχείο αυτό το οποίο ε, αποκαλούν οι Αμερικανοί ε, ότι έχει τα πάντα. δηλαδή καλύπτει μια μεγάλη σειρά θεμάτων που αφορούν την ελευθερία του τύπου και αυτό ε, θα μπορέσει κανείς να πει ότι αυτό αποτελεί επίτευγμα και αυτές είναι οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως μερικές φορές πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω αν έχουν, ε, το γνωρίζουν οι συνάδελφοι, αλλά στο ΕΒ Βασίλειο αυτή τη στιγμή γίνεται μια εκτεταμένη συζήτηση στο Κοινοβούλιο ε, και στην κοινωνία για την ελευθερία του τύπου. Μετά από όλα όσα γίνονται στα μέσα ενημέρωσης, όπου έχουν υποθεί πράγματα για ανθρώπους που είναι διάσημοι στο πολιτικό ή στο μη πολιτικό χώρο και που αργότερα βρέθηκαν στα δικαστήρια ή που έχει αποδειχθεί ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι ένοχοι για ψεύδι ή αν όχι για στρέβλωση και παραποίηση γεγονότων. Υπό τις συνθήκες αυτές υπάρχουν λόγια ανησυχία, Παραδείγματο χάρη, η αστυνομία έχει κυκλοφορήσει πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης για ή και για απλού ανθρώπους με τρόπο που δεν εγκρίνει η κοινή γνώμη. Άρα η πίεση της κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ελευθερία του τύπου είναι μάλλον εχθρική. Και ο ο υπεύθυνος λόρδος που έχει αναλάβει την ε, ε, έρευνα αυτή και έχει έρθει σε επαφή με όλα τα στρώματα της Βρετανικής κοινωνίας, έχει δει ότι υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Για πρώτη φορά στη Βρετανία πρέπει να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα και όχι με τα γενικά. Και στους Times του Λονδίνου διάβαζα σήμερα ότι λέει γιατί αυτοί που ε, γράφουν στον τύπο θα πρέπει να έχουν περισσότερη ελευθερία από τον οποιοδήποτε άλλο στην καθημερινή ζωή. Πολύ ωραίο ερώτημα. Το θεωρούμε δεδομένο ότι ο τύπος πρέπει να είναι ελεύθερος γιατί ελευθερία του τύπου ίσον ελευθερία του λαού. Βεβαίως. Αλλά γιατί θα πρέπει να είναι πιο ελεύθερος ο τύπος από τους υπολείπους. Αυτή ήταν η ουσία της επιστολής και πραγματικά το πιστεύω αυτό. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η συγγήτρια ήταν πάρα πολύ ευφυής και κάλεψε πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματο χάρη στην, πρώτο, ε, στην πρώτη αναφορά όπου αναγνωρίζει ότι οι κυβερνήσεις είναι κυρίως υπεύθυνες για, τον, για το ότι περιορίζεται η ελευθερία του τύπου. Ακριβώς περί αυτού κατηγορείται ο, προ, ο, Πρωθυπουργό και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ε, σήμερα, ότι ε, απειλούν ότι θα περιορίσουν τον τύπο με τρόπο που θα ήταν είναι αδιανόητο κανονικά για τον Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πώ λειτουργούν όλα αυτά. Θα έλεγα στην εισηγήτρια ότι δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι συμφωνώ με τους προλαλήσαντες για το γεγονός ότι δεν, είμαστε συγκεκρι... δεν αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε κάποιες χώρες. Αν θέλουμε να έχει βάρος, να έχει κύρωση η έκθεση αυτή και της αξίζει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχει ένα παράρτημα όπως κάνει κάθε χρόνο η Διεθνής Αμνηστία που φτιάχνει έναν κατάλογο για την κατάσταση της ελευθερίας αυτές. Ίσως θα πρέπει να γίνει και αυτό. Δηλαδή να αναφέρουμε τον κατάλογο των χωρών όπου θεωρούμε ότι η ελευθερία που έχει ο τύπος για τη λειτουργία του δεν είναι τόσο σοβαρή, σημαντική όσο λέγαμε. Έχοντας υπόψη αυτό που είπα ότι στη Βρετανία διαρωτόμαστε αν είμαστε, εμεί αν είμαστε εμείς ελεύθεροι, έχουμε ελεύθερη του τύπου. Το θέτω όμως ρητορικά, γιατί αντιλαμβάνομαι ε, την πρακτική δυσκολία του να πει κανείς για 189 χώρες αν είναι καλές, κακές ή και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο όμως με ανησυχεί και το οποίο ε, ε, προέκυψε επανειλημμένο στη Βρετανία, αυτός ο Λόρδος Λέβισον έχει σχολιάσει ασχοληθεί δεν έχει μπει στα θέματα της ουσίας, τα, ε, τα προσωπικά και το blogging. Τα ψηφιακά μέσα δεν προέρχονται από μια χώρα εξορισμού. Δεν είναι ε, τυπωμένη εφημερίδα στην Κοπενχάγη, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Είναι προέρχονται από κάπου που πολύ συχνά δεν ξέρουμε πού είναι αυτό και δύσκολα ελέγχονται. Και παρότι η εισηγήτρια ε, εξηγεί πολύ σωστά ορισμένα πράγματα, διερωτώ με αν δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε τα συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή το πώς θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Αυτό σαφώς είναι το μεγαλύτερο κοινοβούλιο ελεύθερων κρατών του κόσμου. Και έτσι αυτό ε, μας αφορά, γιατί εμείς έχουμε κράτη-μέλη μεταξύ μας που πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν ελευθερία του τύπου, δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν, Πρέπει λοιπόν να αναγκαστούμε να διατυπώσουμε τη θέση μας. Είναι μια εξαιρετική αρχή. Θέλω να συγχαρώ μέσω εσάς κύριε Πρόεδρε την ε, εισηγήτρια, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το λίγο παραπάνω και να προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι και να το ε, θέσουμε ως κριτήριο για να κρίνονται άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Επόμενος και τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Λαντσβέργης. Ε, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ την κυρία Σχάκε, την εισηγήτρια. Και εγώ θα ήθελα να προτείνω επίσης, όπως και ο Σεράτκινς, να ε, διευρυνθεί ενδεχομένως η έκθεση και να συμπληρωθεί από κάποια σημεία τα οποία θα μου επιτρέψετε να σας πω. Βεβαίως, ποτέ ένα έγγραφο δεν είναι πλήρες. Μπορεί ο καθένας να κάνει τροπολογίες για να το συμπληρώσει, ε, αλλά συχνά η ίδια η συγγήτρια δίνει προσοχή και τα συμπληρώνει από μόνη της. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου, καθώς διαβάζω το κείμενο, είναι το εξής η σχέση μεταξύ των μέσων επικοινωνίας και της ε, ε, βιομηχανίας διασκέδες και ψυχαγωγίες. Αυτό προσπαθεί να δώσει ένα μανδύα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Αυτό όμως τι είναι, είναι μέσο επικοινωνίας, είναι μια βιομηχανία διασκέδασης, business δηλαδή. Είναι μια διάκριση που αξίζει να παρουσιαστεί ή να υπογραμμιστεί με κάποιο τρόπο να αναφέρεται στην έκθεση. Κάποια σχόλια ακόμα για την ελευθερία της έκφρασης. Είναι άρα και πραγματικά ελεύθερη έκφραση και μπορεί να είναι από ένα μέσο ενημέρωση που έχει επιχειρηματικά συμφέροντα. Και είναι ελεύθερο για τους δημοσιογράφους. Όταν ε, ε, είναι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία εμπορική που έχει συμφέροντα, ε, να έχει κέρδη. Δηλαδή είναι ελεύθεροι από κάθε είδους δεσμούς και σχέση υποταγής σε οποιοδήποτε ιδιοκτήτη μέσω ενημέρωσης. Πολύ συχνά αυτό οδηγεί σε ε, εσωτερική ε, λογοκρισία, όχι κρατική, καταλαβαίνετε. Ε, αυτό κάπως θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα τέτοιο επίπεδο όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα έγγραφά του. Τώρα, τι γίνεται με τις ελευθερίες και τους κινδύνους που ενέχουν και πότε κινδυνεύουν. Ορισμένα σημεία που λέτε είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, αλλά πρόσφατα έχουμε δει και περισσότερα περιστατικά. Όταν εκφράζεται πολιτική κριτική ε, στα μέσα ενημέρωσης και πολλές φορές αυτό στιγματίζεται ε, και του βάζουν μια ταμπέλα ή ακόμα και ποινικοποιείται ως υποδάβληση του μίσους. Μα πού είναι η ε, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα ε, στην υποδάβληση του μίσους και την κριτική προς την εξουσία ας πούμε πρώην νομοθεσία για τον εξτρεμισμό στη Ρωσία και όλα αυτά, οποιοδήποτε ε, τολμάει να επικρίνει την κυβέρνηση, ε, ποινικοποιείται και χαρακτηρίζεται εξτρεμιστής, ακραίος. Έρχομαι τώρα στην παράγραφο 9, σε αυτά που λέτε εκεί, ότι χρησιμοποιούνται τα μέσα επικοινωνίας ως κλασικά εργαλεία προπαγάνδας. Δεν είναι μόνο Πολύ ήπια το λέτε εκεί. Τι γίνεται όταν ε, παρερμηνεύονται οι ελευθερίες. Ας πούμε, κάποιοι δημοσιογράφοι ή δημοσιογραφία γενικά ενέχεται, διαπλέκεται ε, ή ε, δωροδοκείται ακριβώς με σκοπό τη δυσφήμιση, τη συκοφάντηση, τη βλασφημία, ε, με σκοπό και πάλι επιχειρηματικά συμφέροντα και χρησιμοποιείται ως δημοσιογραφία πολύ συχνά. Ανισχούμε πάρα πολύ ορισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Σε mi posso permettere personale. Και μια προσωπική παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά την ε, παρέμβαση του συναδέλφου Άτκινς. Συμφωνούμε με την ιδέα ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια, ένας κατάλογος των ανυπότακτων ας πούμε έτσι χωρών, των λιγότερο καλά συμμορφούμενων. Ε, όμως δεν είναι εύκολο να εντοπίσουμε ε, σύνολα, ομάδες προσώπων ε, που να είναι απαρκώς αντικειμενικοί, αδια, αδιάβλητοι τελείως από οποιονδήποτε, ώστε να καταρτήσουν ένα τέτοιο κατάλογο θα μπορούσε να θεωρηθεί μέσω πολιτικής προπαγάνδας, πολιτικής ε, επιρροής ένας τέτοιος κατάλογος. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Και τώρα για τα τελικά τη σχόλια λόγω στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές αλλά και τους υπολείπους οι οποίοι έκαναν σχόλια. Τα εκτιμώ τα σχόλιά σας, δεδομένου ότι ο χώρος που διατίθεται για αυτές τις εκθέσεις είναι περιορισμένος. Υποθέτω ότι οι τροπολογίες θα προσφέρουν μεγάλη ε, προστιθέμενη αξία και θα ξεπεράσουμε αυτά όλα τα, τη γενικότητα των θεμάτων ώστε η κυρία Γιακονσάρη και τον κύριο Άτκινς. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ήμουν εισηγήτρια και για τη στρατηγική της ψηφιακής ελευθερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική της δράση και ελπίζω και πιστεύω ότι κάποια από τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την ψηφιοποίηση ε, για τον μέσον μέσων ενημέρωση, αλλά και πέρα από αυτά έχουν ε, αντιμετωπιστεί στην έκθεση αυτή. Αν όχι, αυτό θα γίνει τώρα. Πάντως σκόπευα να μην επαναλάβω μια σχετικά πρόσφατη έκθεση γιατί ε, τα θέματα της ελευθερίας του τύπου ε, συγκεκριμένα χρειάζονται περισσότερο χώρο από ό,τι ε, διατίθεται σε μια τέτοια έκθεση. Αλλά όσο μπορούμε να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες φυσικά τόσο το καλύτερο. Τώρα, ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ, θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να ε, αναφερθεί συγκεκριμένα. Καμιά φορά όμως διστάζω να μιλάμε στον, για τον εαυτό μας γιατί έχουμε την ικανότητα να βελτιώνουμε τις λειτουργίες μας μέσω των αντιπροστιψιών μας με τις αναφορές, διαπραγματεύσεις, συμφωνίες που κάνουμε και μέσω της, των αναφορών που υποβάλλουν στο Κοινοβούλιο αυτό η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως θα πρέπει αυτό να το διατυπώσουμε πιο ξεκάθαρα και έχει νόημα. Ευχαριστώ την κυρία Γιακονσάρη. Επίσης άκουσα αυτό που προτείνετε για το θέμα του, να είμαστε συγκεκριμένοι για το θέμα της ιδιοκτησίας και του προλαραλισμού. Θα το κάνω. Δεύτερον, όσον αφορά το, το θέμα των συγκεκριμένων χωρών, την αναφορέ σε χώρε, αυτό είναι συγκεκριμένο δίλημα. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ούτε, ούτε μία χώρα που δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Εγώ είμαι Ολλανδή, είναι γνωστή μια ως φιλελεύθερη και ελεύθερη χώρα όπου η ελευθερία του, της έκφρασης χαίρει μεγάλη εκτίμηση αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα για τους δημοσιογράφους και για το θέμα της ψηφιοποίησης. Σαφώς παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο Ενωμένο Βασίλειο αποτελεί την έμπνευση του σημείου 20 όπου αναφέρεται ότι πρόσφατα κάποια μέσα ενημέρωσης ε, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστεί έλεγχο για την ε, ιδεολογική του συμπεριφορά και ότι θα πρέπει να μπορούμε να διδάσκουμε όταν και εμείς είμαστε εντάξει. Επίσης επισημαίνω ότι πιστεύω ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δυσκολίες που υπήρχαν στο, στις περισσότερα κράτη-μέλη και στις ε, καταστάσεις ζωής ή θανάτου που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι και κάποια μέσα ενημέρωση σε τρίτες χώρες. Άρα σαφώς αναγνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη μας, όμως νομίζω ότι αυτές δεν συγκρίνονται ε, ώστε λοιπόν για να ανταποκριθώ στις προτάσεις ε, της δικές σας κύριε Πρόεδρε γιατί να μην κάνουμε ε, μια πρόταση για ένα παράρτημα το οποίο να έχει διάφορους καταλόγους που ήδη συντάσσουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις κάθε χρόνο, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα μεταξύ άλλων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων επίσης κάνει μια κατάταξη κάθε χρόνο και επίσης γνωρίζουμε το Freedom House, Freedom of the Press, τις εκθέσεις τους. Ε, αυτές είναι τρεις οργανώσεις, υπάρχουν και άλλες. Θα μπορούσαμε να συντάξουμε λοιπόν ένα, μια σειρά καταλόγων, μια σειρά από κατατάξεις ώστε να μην μπούμε στη δύσκολη θέση να αξιολογήσουμε εμείς τι είναι σωστό και τι δεν είναι που θεωρώ δυστυχώς ότι θα, θα περάσει σε συζήτηση μετά θα, γιατί κάποιοι προτιμούν κάποιες χώρες και άλλοι τις επικρίνουν. Έτσι, ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση. Ελπίζω με τους ε, σκιώδεις να το συζητήσουμε. Προ τον κύριο Λατσμπέργκης τώρα αυτά που είπατε για την χειραγώγηση των ε, μέσων ενημέρωσης για να αντιμετωπιστεί η διαφωνία, η, τα διαφωνούντα μέσα ενημέρωσης ή κυρίως για να χρησιμοποιηθεί η κοινή γνώμη ε, ώστε η οποία μπορεί να στραφεί κατά αυτών που επικρίνουν κάποιους, είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίσης αναφερθήκατε στη διάκριση μεταξύ της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης και καμιά φορά ε, το επιχείρημα ότι τα ελεύθερα, ε, τα, ε, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιείται για να, να νομιμοποιηθεί συμπεριφορά που δεν θα έπρεπε να νομιμοποιείται. Υπάρχουν πράγματι ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Εγώ πιστεύω ότι προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Είναι όμως μια φιλοδοξία την οποία θα πρέπει να επιδιώξουμε. Ε, αυτό κάνουμε με την έκθεση αυτή. Επίσης αναφερθήκατε στην δυσκολία της ε, διάκρισης του πολιτικού λόγου σε σχέση με τον εξτρεμισμό. Αυτό το ανέφερα με το θέμα της, ε, του εισηκοφάντησης, ε, της χρήσης των αντιτρομοκρατικών νόμων κλπ. Αλλά αν θέλετε μπορώ να κάνω πιο συγκεκριμένες αναφορές αν ε, ακούω όλα τα σχόλια και με τα μεγάλης χαράς διαπιστώνω ότι υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και προσβλέπω στη συνεργασία μου με τους ε, σκιώδεις και οποιονδήποτε άλλο θα ήθελε να υποβάλει τροπολογίες. Και ε, επίσης σχετικά με το ψηφιακό σκέλος, δείτε την έκθεση ε, την προηγούμενη για την, την ψηφιακή στρατηγική. Επίσης η κυρία Γιάκονσεν ταυτόχρονα αναφέρει για μια, μια έκθεση που συντάσσεται στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και αυτά τα λέω για να ε, μην κάνουμε επαναλήψεις και επικαλύψεις και να καλύψουμε και τα θέματα που δεν εμπίπτουν στις δύο αυτές εκθέσεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόθεση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης. συγητής, Φρανσίσκο Χωσέ Μιλάν Μον, η πρώτη εξέταση μιας έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίες για, σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, και την πρόθεση της ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης. Θέλω να υπενθυμίσω στην ε, Επιτροπή ότι το Διευρυμένο Προεδρείο αποφάσισε η έκθεση αυτή να ε, έχει δύο στόχους. Πρώτον, της διμερείς σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα ΕΕ, υπό το φως της δεύτερης θητείας του Πρόεδρου Ομπάμα και δεύτερον το πλαίσιο αυτών των σχέσεων σε μια ευρύτερη διατλαντική συνεργασία που συμπεριλαμβάνει και τον Νότιο Ατλαντικό και που ανοίγει νέες δυνατότητες συνεργασίας με χώρες Λατινικής Αμερικής. Δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη από τον περασμένο μήνα Είχα την ευκαιρία να κάνω μια πρώτη παρουσίαση της έκθεσης αυτής βάσει ενός εγγράφου εργασίας που τότε σας είχε διανεμηθεί. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να επαναλάβω όλα αυτά που είπα τότε. Το είπατε κι εσείς, Πρόεδρε, πολύ ωραία. Διπλή ήταν η εντολή μου. Πρώτον, η κλασική, ας πούμε, διατλαντική σχέση μετά την επανεκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα και κατά δεύτερο λόγο, ακριβώς να δούμε μια ευρύτερη ατλαντική προοπτική που θα συμπεριλάβει όλο το χώρο του Ατλαντικού, για να το πω έτσι. Θα ήθελα να πω ότι είναι δύο ε, ξεχωριστά τμήματα, δύο ενότητες, οπότε και η έκθεση είναι περίπου δυτή. Ε, παρόλο που ήσασταν γενναιόδοροι μαζί μου. Είναι, έχω περιορισμό από τους κανόνες του Κοινοβουλίου για την έκθεση πρωτοβουλίας σε αριθμό χαρακτήρων και σελίδων. Πρώτον, σχέση λοιπόν Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα που εξελέγει ο πρόεδρος Ομπάμα, υπάρχει ευκαιρία να α, δώσουμε μια νέα πνοή στις σχέσεις μας. Παρόλο που λέγουν ορισμένοι ότι στρέφεται η Αμερική προς τον ειρηνικό ε, όχι μόνο από την εκλογή του Ομπάμα, αλλά και γενικότερα ε, με την προοπτική διαπραγμάτευσης για μια συμφωνία ε, εταιρικής σχέσης, εμπορικής και επενδύσεων. Αυτές οι διαπραγματεύσεις και η τελική σύναψη της συμφωνίας νομίζω θα άνοιγαν ένα πεδίο συνεργασίας και πέρα από το διμερές Ε, θα έχουμε νέα πρότυπα για τις δημόσιες προμήθειες, για την πνευματική ιδιοκτησία, πρότυπα κτλ. Υπάρχουν ε, μεγάλες χώρες πλέον που είναι οικονομίες ε, παγκόσμιες, η Κίνα κτλ. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να αναζωογονηθεί η σχέση μας και να δείξουμε και στον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν φθήνει, ότι είναι ζωντανή, στεναρή, φιλόδοξη ε, και στραμμένη προς τον παγκόσμιο κόσμο και την παγκόσμια οικονομία και δεν θέλουμε να έχουμε ένα ρόλο έτσι περιθωριοποιημένο. Αυτά ποσοτικά Καταλαβαίνουν, καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο κείμενο στην έκθεσή μου. Ένα ψήφισμα που ενέκρινε η ΙΝΤΑ, η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, τον Οκτώβριο, είναι σχετικό και σήμερα ήμουν σε αυτή την Επιτροπή και πάλι ετοιμάζουν δικό τους ξεχωριστό ψήφισμα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε ήδη, ε, δίνω ε, μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα, αλλά όχι μεγάλο όγκο στην έκθεσή μου, γιατί έχω περιορισμό και μιλώ επίσης για την εξωτερική δράση στον παγκόσμιο αυτό κόσμο που ζούμε, ότι χρειάζεται να είναι συντονισμένη. Ε, η εν τι ενώση, προφανώς, και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να συντονιστούν όσο γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για παγκόσμιες προκλήσεις, αλλά και για περιφερειακά ζητήματα σειράξης ε, Συρία, Αφγανιστάν, ε, Κίνα, Ρωσία, ε, η Αραβική Άνοιξη. Πάντα μιλώ λοιπόν για συντονισμό και συνεργασία. Υπό την έννοια αυτή επαναλαμβάνω κάτι που πάγια έχει πει το Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα, ότι είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα είδος πολιτικού διατλαντικού συμβουλίου. Και εκεί να είναι ο κύριος Κέρι, η κυρία Άστον ή ο, ο διάδοχός της και κάθε τρίμηνο ας πούμε να ε, αναφέρουν για ζητήματα τέτοια προκλήσεις εξωτερικής πολιτικής γιατί όχι και καμιά φορά καμιά στρατηγική ανάλυση. Επίσης, ε, ο διατλαντικός διάλογος ε, των νομοθετών ανοίξαμε γραφείο στην Ουάσιγκτον και θα θέλαμε και το Κογκρέσο να ανταποδώσει και να ανοίξει εδώ γραφείο. Και επίσης άλλα θέματα δικαιοσύνης εσωτερικών, ανταλλαγή δεδομένων, καταπολέμηση της ομοκρατίας, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά είναι θέματα ε, που έχουμε και κοινή ε, συνεργασία το 2010, το θέμα των θεωρήσεων για τέσσερα κράτη-μέλη ε, κρεμεί ακόμα, δηλαδή οι πολίτες από τέσσερα κράτη-μέλη χρειάζονται βίζα για να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έρχομαι τώρα στην παγκόσμια προοπτική, στο δεύτερο τμήμα της έκθεσής μου. Όπως σας είπα, ξέρετε ότι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες. Στο German Marshall Fund έχουν γίνει ενδιαφέρουσε μελέτες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 ε, και ένα συμπόσιο έγινε για τις προκλήσεις σε θέματα ασφαλείας ε, από το 2011 ένα σεμινάριο μέχρι η κυβέρνηση του Μαρόκου εργάζεται προς την κατάσταση αυτή. Ε, το 2009 έγινε μια διάσκεψη, μιλούν για μια διατλαντική κοινότητα εκείνη ε, και γενικά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια επιθυμία για μια εταιρική σχέση διατλαντική που απορρέει από το γεγονός ότι έχουμε επίγνωση ότι και οι χώρες που βρέχονται από τον Ατλαντικό θα πρέπει να συνεργάζονται για θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία, παγκόσμια και συνολική, όχι μόνο του Βορρά αλλά και του Νότου. Ε, αναφερθήκαμε στον Ειρηνικό και στην Ασία. Αφού λοιπόν γίνεται τόσο λόγο για τον Ειρηνικό, γιατί εμεί να μην στραφούμε στον Ατλαντικό και προ τον Νότιο Ατλαντικό, Βραζιλία, Μεξικό και λίγο πιο πάνω. Αλλά και στην Αφρική χώρε όπω είναι η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, αυξάνεται η ενεργειακή παραγωγή στι χώρε κεντρική ε, ε, Αφρικής, ε, Δυτικής Αφρικής κτλ. Και μετά γίνεται ειδικό λόγος για τη δίσδυση της Κίνας και στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Αυτό ίσως εξέπληξε τις χώρες του Βορρά που θεωρούσαν ότι παραδοσιακά ήταν παρούσες οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη και τώρα έχουν έρθει οι Κινέζοι. Μήπως θα πρέπει να ξαναστρέψουμε εκεί την προσοχή μας. Όχι μόνο στο Βόρειο Ατλαντικό, αλλά και στο Νότιο Ατλαντικό. Έπαιξε και αυτό ρόλο. Λοιπόν, στην έκθεσή μου εγώ κάποιες προτάσεις κάνω και τίποτα παραπάνω ποιοι είναι οι φορείς με τους οποίους θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ένωση να σκεφτούν με ποιους συνομιλούμε και ε, σας είπα προηγουμένως ήδη χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουμε πολλές κοινέ αξίες, αρχές, οράματα, ακόμα και την εικόνα που έχουμε για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Είναι οικονομίες της αγοράς ελεύθερες με κάποιες ε, εξαιρέσεις να έχουμε ένα τριμερή διάλογο Τώρα στην ουσία, στην πράξη λίγα πράγματα συμβαίνουν, αλλά ε, οι θεσμοί υπάρχουν. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Βέβαια η Λατινική Αμερική είναι ετερογενής, δεν είναι ομοιογενής. Υπάρχουν πολλές περιφερειακές ενώσεις, ΣΕΛΑ, Κονασούρ και διάφορες άλλες υποπεριφερειακές που θα υπήρχε προστιθέμενη αξία στην παγκόσμια διακυβέρνηση, στην κλιματική αλλαγή, πολύ σημαντική εκεί, στο θέμα της εγκληματικότητας, άλλο σημαντικό θέμα για την περιφέρεια, και οικονομικά και εμπορικά. Εάν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ και με τον Καναδά, θα βρεθούμε στην επόμενη φάση. Έχουμε συμφωνίες με το Μεξικό, την Κίνα, την Χιλή, συγγνώμη, το Περού και την Κολομβία, ελευθέρων συναλλαγών και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αντίστοιχες συμφωνίες με τις ίδιες χώρε. Κεντρική Αμερική, Περού, Κολομβία, Χιλή και εκτός ε, από την, αυτά, απ' την άλλη υπάρχει με το Μεξικό και ε, τον Καναδά. Λοιπόν, αν όλα αυτά στεφτούν με επιτυχία θα έχουμε ένα τεράστιο τρίγωνο με αυτές τις χώρες και μπορεί να τελειώσουν και οι διαπραγματεύσεις κάποτε με τη Μερκοσούρ. Λοιπόν, αυτά όλα είναι τα θέματα που απασχολούν την έκθεσή μου, που μπορεί να έχουν τη αξία. Σας είπα για την παγκόσμια διακυβέρνηση, με ποιους μηχανισμούς. Είπαμε ποιες είναι οργανώσεις που υπάρχουν και ε, η Συμμαχία για τον Ειρηνικό, Καρικό. Υπάρχουν διάφοροι περιφερειακοί οργανισμοί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να υπάρχει τριγωνική συνεργασία, ρεαλιστική, επιμέρους, σταδιακή, βαθμιά, ανάλογα με τους εταίρους μας. Έχουμε με τη ΣΕΛΑΚ ε, αναδιετία ε, Σύνοδο Κορυφής. Η δικιά μας θα είναι το 2015 με τις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης το 2015 στον Παναμά. Ε, θα μπορούσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις για τις Συνόδους Κορυφής που έχουμε με τις Λατινοαμερικανικές χώρες, κάθε Και μουτά της Μπουτάντης υπάρχει και η άλλη πλευρά, ε, η Αφρική, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στην Αφρική και οι προκλήσεις που έχουμε είναι παγκόσμιες, ναρκωτικά ασφάλεια είναι γνωστό άλλωστε ότι το θέμα αυτό δεν είναι μόνο τριγωνικό πλέον, αλλά τετράγωνο. Η κοκαίνη πηγαίνει από τη Λατινική Αμερική προς Βορράν, ε, Μεξικό, Ηνωμένε Πολιτείε και άλλη προς τη Δυτική Αφρική και από εκεί ε, ανεβαίνει στην Ευρώπη. Δεν είναι τρίγωνο πλέον, έχει γίνει τετράγωνο αυτή η ιστορία ε, των ναρκωτικών. Και θα ήταν πολύ χρήσιμο να συνεργαστούμε εκεί στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, η διακίνηση, του λαθρεμπόριου όπλων και όλα αυτά είναι θέματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τετραμερούς πλέον διαλόγου. Επίσης, πειρατεία, άλλο θέμα. Και υπάρχουν βοήθειες οικονομικές ε, και από τη ΣΥΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Οικονομική Οργάνωση Δυτικής Αφρικής, ΣΕΝΤΕΑΟ, και ε, άλλη περιφερειακή οργάνωση έχουν στην Αφρική με διάφορους οργανισμούς, ακόμα και η ΣΑΝΤΕΚ, που είναι βέβαια ε, στην Μεσημβρινή Αφρική και σε μεγάλο βαθμό προς τον Ινδικό ωκεανό στραμμένη, υπάρχουν μηχανισμοί, μπορούμε να βρούμε και θέματα και ε, επίκαιρα ζητήματα ε, σε τριγωνική σχέση με τη Λατινική Αμερική ή τετράγωνο με την Αφρική. Αυτά. Κάποιες προτάσεις κάνω. Δεν θέλω να φτιάξω δόγμα ε, σε ένα θέμα τόσο περίπλοκο και τόσο δύσκολο. Τελειώνω, Πρόεδρε, τελειώνω. Σήμερα επίσης δεν πιστεύω ότι κατά κύριο λόγο κυριαρχεί αυτό το θέμα στις χώρες αυτές πιο πολύ σκέφτονται τους τοπικούς οργανισμούς παρά τις παγκόσμιες ε, συνεργασίες αλλά πολλοί όμιλοι προβληματισμού think tank έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα για να έχουμε μια κοινή συναντήληψη για μια κοινότητα του Ατλαντικού που να συμμετέχουν όλες αυτές οι χώρες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, θέλω να ακούσω και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αλαφράγκα. Όχι. Κυρία Νέτ, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σαλαφράγκα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μιλανμόν για την έκθεση αυτή, η οποία είναι διεξοδική είναι τόσο διεξοδική γιατί προσπαθεί να καλύψει κάθε πτυχή της διεθνούς πολιτικής αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά κανείς να κάνει μια επιλογή. Καλό λοιπόν θα ήταν να επιχειρήσουμε να επικεντρωθούμε σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς κατόπιν επιλογής. Και ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη φάση είναι οι διαπραγματεύσει για τις εμπορικές συμφωνίες, για την εμπορική συμφωνία συγκεκριμένα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν οι δύο πλευρές συμφωνούν για τους γενικότερους, απότερου στόχου, το να επεξεργαστούμε τι λεπτομέρειε θα είναι και πολύ δύσκολο και θα μα Θα είναι μια πραγματική πρόκληση για μια σειρά από λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί ο στόχος δεν είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ως αυτό σκοπό. Πρέπει να κάνουμε σωστή διάκριση μεταξύ και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, να συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερομένους, ξεκινώντας με τους βουλευτές εδώ στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την γεωργία θα έχουν άλλη σκοπιά προφανώ για τι εμπορικέ σχέσει με τι ΗΠΑ από ότι συνάδελφοι που ενδεχομένω ενδιαφέρονται περισσότερο για την ψηφιοποίηση, τη βιομηχανική πολιτική και ούτω καθεξής. Αυτό θα είχα να συστήσω. Και έπειτα, όταν ζητούμε νέα σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων τότε καλό θα ήταν να καλέσουμε τα κρατημέλη να αποφύγουν τα σφάλματα του παρελθόντος Δηλαδή, ήταν πολλοί οι Ευρωπαίοι συμμετέχοντες που ήθελαν να έχουν χρόνο ομιλίας, αλλά έτσι υποχρεώθηκαν οι Αμερικανοί ε, συμμετέχοντες να περιοριστούν σε μια σειρά από πολύ σύντομε παρεμβάσει, χωρί ιδιαίτερο νόημα. Βαρέθηκαν οι Αμερικανοί και δεν κατάλαβαν και τι γινόταν τελικά. Για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Προ δικό μας όφελος λοιπόν θα είναι να το προβλέψουμε αυτό στο μέλλον, να το προλάβουμε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά θυμάμαι κιόλα ότι στην εκπόνηση προηγούμενων εκθέσεων, νομίζω πέρυσι πριν δύο χρόνια, κάποιες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου είχαν επισκεφτεί το Κογκρέσο στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και μάλιστα, επί δυόμιση μήνες πήγαιναν και ξαναπήγαιναν. Ήταν κουραστικό. Και παραξενευτήκαμε που δυσκολευόμασταν να συναντήσουμε του Αμερικανού ομολόγου. Μα αν έπρεπε να συναντούν τον καθένα, την κάθε μια αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πέρασε από το Κογκρέσο, κάποιοι δεν θα είχαν χρόνο να κάνουν τίποτα άλλο στη ζωή του. Πρέπει λοιπόν να γίνει κι άλλη δουλειά. Πρέπει οι σχέσει μα να γίνουν αποτελεσματικότερε. Απευθύνω έκκληση προ του συναδέλφου και προ όλου να την κάνουμε την προσπάθεια αυτή. Κατανοώ πλήρω ότι δεν είναι απλό το εγχείρημα. Αλλά να προσπαθήσουμε πραγματικά. Απευθύνω έκκληση προς όλους, όλους μας. Να διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα, να διευκολύνουμε την άναξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελεύθερου Μπορείου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, των ε, Μιλάν Μον, για τη δουλειά του. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και παραδέχομαι ότι έχω κατανόηση. Ενδεχομένως μερικές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο ευρύτερα και να ξεπερνάμε τα όρια της καθημερινής ε, ρουτίνας και δουλειάς. Όμως, ε, συμφωνώ και με αυτά που είπε η κυρία Νέιτς, ότι θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε ε, σε θέματα προτεραιότητας. Έχω κάποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να είναι μέρη τροπολογίες στην έκθεσή σας ε, και κάποιες άλλες να τις περιμένετε. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρία θέματα. Πέρα από το θέμα του εμπορίου και των επενδύσεων θα πρέπει να επικεντρωθούμε από κοινού σε κάποια άλλα. Το ένα είναι το θέμα του κλίματος. Ο πρόεδρος Ομπάμα στην εναρκτήρια ομιλία του ε, ε, ανέφερε όπως και σε άλλες ομιλίες ότι θέλει τη δεύτερη θητεία του να τη χρησιμοποιήσει για να ασχοληθεί πρακτικά με αυτό το ζήτημα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να, ε, να διστάσουμε να πιστέψουμε αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Αυτό πρέπει να είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει γιατί πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Δεύτερον, εγώ θα ήθελα να μιλάμε πιο ξεκάθαρα για τη Μέση Ανατολή πιο ξεκάθαρα από ό,τι μέχρι τώρα να ε, χρησιμοποιεί η έκθεση, γιατί κατά την άποψή μου αυτό θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικότερη προτεραιότητα και αυτό πρέπει να διαφανεί. Τρίτον, επίσης θα ήθελα να δοθεί περισσότερη έμφαση στο ζήτημα του αφοπλισμού και στο ζήτημα της ασφάλειας. Όχι μόνο δηλαδή να περιγράφουμε τις δυσκολίες, αλλά να χρησιμοποιούμε τις ευκαιρίες αυτές για να καταλήξουμε και εμείς σε συμπεράσματα. Μια τελευταία παρατήρηση. Είναι πάντοτε δύσκολη, λο να προτείνει κανείς τη δημιουργία ενός οργάνου, ενός θεσμικού οργάνου, μιας διάσκεψης κορυφής, μιας νέας οποιασδήποτε νέας δομής. Αν όμως ε, αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα την ενισχυμένη συνεργασία στην οποία στοχεύουμε, τότε θα έχουμε πρόβλημα της ε, δημοκρατικής νομιμοποίησης της διατλαντικής σχέσης. Γιατί πάρτε το παράδειγμα των διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που θα έχει συναυθεί η συνθήκη, ποιος θα είναι ο υπεύθυνος, το υπεύθυνο όργανο που θα, επαν, θα εξετάσει τυχόν αλλαγές και που θα έχει δημοκρατική νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο. Όταν δημιουργήσαμε κοινή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα δημιουργήσαμε ένα κοινοβούλιο για να επιβλέπει την κοινή αγορά. Τώρα που δημιουργούμε κοινή αγορά με τους Αμερικανούς, ποιο θα είναι το αντίστοιχο μέτρο που θα ε, δημιουργήσει την, ε, που θα δώσει την νομι, ε, δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτή είναι μια ιδέα που θα ήθελα να τη συζητήσουμε. Κύριε Σαλαφράγκα, Κύριε παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Μιγιάν για την έκθεση αυτή που έχει ως επικεφαλίδα ο ρόλο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόθεση μια ευρύτερη διατλαντικής εταιρική σχέση. Ο κύριος Μιγιάν, όπως πάντα, είναι πάρα πολύ επιμελής και συστηματικός στην προσέγγιση του και μέγας γνώστης, όπως απέδειξε. Και το έχει αποδείξει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ε, στον διατλαντικό νομοθετικό διάλογο. Δεν με ε, εκπλήσει αυτό που προτείνει ο κύριος Μπουτικόφερ είναι πράσινος μεν, αλλά λαμπρός ε, εκπρόσωπος των πρασίνων, όχι ο μόνος. Ε, είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή και πάρα πολύ επίκαιρη η έκθεση γιατί όλες οι μελέτες, όλες οι αναλύσεις ε, προοπτικής δείχνουν ότι μέχρι το 2035 ο παγκόσμιος οικονομικός άξονας θα έχει περάσει από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό και Ινδικό ωκεανό. Οπότε, τι λέμε με την έκθεση αυτή, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει σημαντικά ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, η, η μόνη υπερδύναμη δεν είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι αποφάσεις δεν παίρνονται στον κόσμο από το G8, ε, δεν κυριαρχούν εκεί αυτές οι δυνάμεις. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να βαθύνουμε σε ένα διάλογο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν να προσφέρουν πολλά ακόμα. Βλέπουμε τα στοιχεία των επενδύσεων, το παγκόσμιο ΑΕΠ, τις συναλλαγές. Ε, είναι δύο πρωταγωνιστές εκ των ΟΚ άνευ. Θα ήθελα λοιπόν να πω εδώ, Πρόεδρε, ότι η έκθεση αυτή συνδυάζει δύο πάρα πολύ εύστοχα στοιχεία. Πρώτον, γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις. Ο κύριος Μπιουτικόφερ ε, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα και θα σηκώσω το γάντι και εγώ και θα ε, το υποβάλω στον εισηγητή να εμβαθύνει στην ιδέα αυτή. Τι μας ζητάει, να έρθει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ολομέλεια να ε, γίνει μια σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για να δούμε μέσο και μάκρο πρόθεσμα αλλά και βράχει πρόθεσμα τα διμερεί και τα παγκόσμια θέματα και ο κύριος Μπιτικόφερ μιλάει και για μια δημοκρατική νομιμότητα ε, στα θέματα που μας απασχολούν. Μα κύριε Μπουτικόφερ, αυτό τον καιρό Έχουμε μια ισομερή συνέλευση ΑΚΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την Ευρωμεσογειακή Συνέλευση, έχουμε Ευρωλατινοαμερικανική Συνέλευση και έχουμε και Euronest με τις ε, χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και της Βόρειας Γειτονίας. Λοιπόν, ε, ζώνη ελευθερών συναλλαγών ε, θέλουμε και να τη γεμίσουμε και με πολιτικό περιεχόμενο, θα μπορούσαμε να έχουμε αντίστοιχη κοινοβουλευτική συνέλευση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αλλά θα ε, το αφήσω στα χέρια του εισηγητή να δει με ποιο τρόπο θα το προσθέσει στην έκθεση του. Συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Πιτικόφερ. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση που αναφέρει ο εισηγητή και δεν θα αντισταθώ στον πειρασμό να το ρωτήσω γιατί ζητάει υπό το φως των συμφωνιών που έχουμε με χώρες Λατινικής Αμερικής, με το Μεξικό κτλ. και με τον Καναδά, να ζητήσουμε, λέει στο σημείο 9, οι δύο εταίροι να μελετήσουν κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια ε, διευρυμένη διατλαντική συνεργασία και στο 10 λέει να προβαίνουν οι εταίροι σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ανταλλαγέ απόψεων σχετικά με τι αντίστοιχε διασκέψει κορυφή με χώρε Λατινική Αμερική. Τώρα, τέτοιε ώρε, τέτοια λόγια. Είναι σκόπιμο να συζητούμε για τριγωνικές συνελεύσεις με την Αμερική. Μήπως είναι πολύ νωρίς. Ίσως όμως πιο μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη αυτή την πρωτοβουλία στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ή σε άλλες διμερείς συναντήσεις που μπορεί να έχουμε. Γιατί νομίζω ότι η παγκόσμια ατζέντα αυτό τον καιρό είναι γεμάτη με θέματα που θα μπορούσαμε να ε, έχουμε μια τέτοια τριγωνική συνεργασία και οι μεγάλες προκλήσεις σίγουρα οι παγκόσμιες εννοώ το ε, δικαιολογούν. Ευχαριστώ τον κύριο Μιγιάν λοιπόν. Ε, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις σε πρωτοβουλία και προοπτική ε, με βάση τις προτεραιότητες και του κυρίου Ομπάμα. Ο κύριος Μπιτικόφερ επίσης προτείνει πέρα από το Ιράν και τα πυρηνικά είναι και η κατάσταση Μέση Ανατολή που μας ε, ενδιαφέρει και ο κύριος Ομπάμα στην αρχή της πρώτης είχε εκφωνήσει μια ομιλία στο Κάιρο δεν ευδοκίμησε αυτή η ιστορία. Έχουμε νέες συνθήκες, έχουμε νέα τοποθέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις και όλο αυτό το θέμα ε, του Αραβικής Άνοιξης έχει μια νέα τακτική είπα, η, εκ των μετόπιστεν ηγεσία leading from behind κάνει λίγο πίσω λοιπόν να δούμε τι θα μας προτείνει ο εισηγητής that the deadline for amendments is the 27 March at noon. Στις 27 Μαρτίου το μεσημέρι λίγη η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Τελευταίος ο μιλητής ο κύριος Λάνθμπεργκ. Έχω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για την πρότασή του Είναι ένα νέο όραμα, διευρυμένο πρέπει να ομολογήσω, για τη διατλαντική σχέση. Η έκθεση, ίσως για πρώτη φορά, δίνει μια νέα φρέσκια αντίληψη, νέα πνοή ε, του ευρωατλαντικού τριγώνου. Πέρα από τη διατλαντική σχέση, που βεβαίως κυριαρχεί και είναι και λογικό, που είναι οι διμερείς σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, υπογραμμίζει προτεραιότητες και συγκεκριμένες δράσεις για τα καθήκοντα του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλην όμως υπάρχει και ένα σημείο ακόμα. Μιλάτε για ένα τρίγωνο που είναι οι δεσμοί μας που είναι η παλιά, η γυραιά, η πυρος, η κουρασμένη Ευρώπη και δύο νεότερες ε, κόρες, θυγατέρες, πολύ δυναμικές και στο ένα πέμπτο της ηλικίας της Ευρώπης που είναι η Βόρεια και η Νότια Αμερική, οι δύο Αμερικές. Εάν λοιπόν αυτό το τρίγωνο μπορεί να γίνει πραγματική συνεργασία και κοινή θέση στον κόσμο σε παγκόσμια κλίμακα πλέον, αυτό θα ήταν μεγάλη ισχύς και μεγάλη ελπίδα επίσης για τον πολιτισμό μας. Αυτό πραγματικά με χαροποιεί πάρα πολύ. Έχουμε δεσμούς ιστορικούς, ε, πολιτιστικούς, κληρονομιά. Ίσως αυτό ε, θα μπορούσατε να το τονίσετε περισσότερο στην αιτιολογική σκέψη ε ή κάπου αλλού. Ε, να το τονίσετε ακόμα περισσότερο είναι πάρα πολύ σημαντικό και νέο στοιχείο. Ευχαριστώ. for answers. Ευχαριστώ. Ας αρχίσω από την κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ κυρία Νέιτς. Πράγματι, η σχέση διατλαντική με τις ΗΠΑ είναι τόσο ευρεία που χρειάζεται να ορίσουμε προτεραιότητες γιατί καλύπτονται όλα τα θέματα. Εμένα δεν μου ζήτησαν μόνο προτεραιότητε. Από την τέσκεψη των Προέδρων μου ζήτησαν να δώσω και μια ευρύτερη προοπτική για το Ατλαντικό γενικότερα και τη διατλαντική σχέση, που ήταν πραγματικά επικίνδυνη αποστολή αυτή. Σχεδόν αδύνατη. Συμφωνώ μαζί σα ότι είναι επίκαιρη τώρα οι σχέσεις. Μιλώ τώρα για βορρά-βορρά, ε, διατλαντική, και κινούν οι διαπραγματεύσεις για την ε, συμφωνία την εμπορική και την επενδυτική. TTIP. Η θέση μου είναι ότι η έκθεση δεν είναι κάτι το αφηρημένο γενικά στο χώρο, αλλά έχει κάποιες αρμοδιότητες μια έκθεση πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο. Σας είπα, σήμερα το πρωί ήμουνα σε συνεδρίαση της ΣΥΝΤΑ, ε, που είχαν την καλοσύνη να μας καλέσουν και εμάς με άλλες επιτροπές, γιατί εκφωνούν για τη συμφωνία αυτή ειδικό ψήφισμα. Και ε, είναι καθήλυνα αρμόδια ή η Επιτροπή αυτή, επί της ουσίας, όπως λέμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Στις 20 τόσο του Οκτωβρίου, δεν θυμάμαι πότε, εγκρίθηκε αυτό το ψήφισμα τους από την Ολομέλεια και δεδομένων των αρμοδιοτήτων που έχουμε εδώ στο Κοινοβούλιο, εγώ δεν μπορούσα να μπω περισσότερο σε λεπτομέρειες. Και σας λέω ότι είναι ένα θέμα που υπερβαίνει την αμυγή οικονομική και εμπορική διάσταση και έχει και τη δυνατότητα ενίσχυσης της σχέσης ε, ε, Ουάσιγκτον-Βρυξελών. Πάρα πολύ. Συσφίγγονται οι δεσμοί. Πολύ περισσότερο. Και υπερβαίνει τα θέματα της επικαιρότητα. Γι' αυτό στο σημείο 3 ή 4 λέγω ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφή θέλω να συζητηθεί αυτό το θέμα, να υπάρχει στην διάταξη αλλά από πλευρά αρμοδιοτήτων δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Για τις συνόδου κορυφής, εγώ έχω πιο αισιόδοξη από εσά άποψη. Είναι ετήσιε οι σύνοδοι κορυφή και θεσμοθετημένε. Δεν είναι τίποτα το έκτακτο, το εξαιρετικό. Πέρσι δεν ε, έγινε λόγω των εκλογών. Αλλά οι σημερινέ σύνοδοι κορυφή από τη συνθήκη τη Ρώμη και μετά είναι πιο ελκυστικέ. Το θέμα τι έγινε με τον Ομπάμα όμω. Το 2009 θυμάστε ήρθε στην Πράγα και ήταν η παλιά μορφή με τους 27 κρατο, ε, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων και η τότε τσεχική κυβέρνηση αν θυμάστε. Δεν θα επεκταθώ. Ε, δεν ήταν πάρα πολύ ελκυστικό αυτό, 27 φωνές, δεν ήταν πάρα πολύ γοητευτικό το σχήμα, ο καθένας είχε τα ζητήματά του, ε, με τη νέα συνθήκη λοιπόν, τη συνθήκη της Λισαβόνας και τα νέα όργανα που έχουμε, που έχουμε ένα μόνιμο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει αλλάξει τελείως το σχήμα προς το καλύτερο. Και δημιουργείται μια, θέση, μια σχέση πλέον εμπιστοσύνης, φιλίας κτλ. Οι σημερινέ συνοδικορυφεί λοιπόν νομίζω θα πρέπει να είναι πιο καλέ, πιο αποτελεσματικέ, πιο ελκυστικέ ε, από τι προηγούμενε, για τι ΗΠΑ ενώ πριν τη Λισαβόνα εποχή. Ε, δεν μπορώ να επικεντρωθώ, δεν μπορώ με την έκθεσή μου να υποκαταστήσω τις αρμοδιότητες της ΣΥΝΤΑ. Για τον κύριο Μπιουτικόφερ, σας ευχαριστώ για τα δώσα καλά σας λόγια και για τη συμπάθεια που δείχνετε, για τις τροπολογίες καλώς να ορίσουν. Ε, θα τις μελετήσω με την αρμόζουσα προσοχή και τη δέωσα. Για την κλιματική αλλαγή λέγεται ότι έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Ομπάμα Μα ορίστε, με τηλεπάθεια έχουμε μεταξύ μας. Το σημείο 22, λέω, ε, επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση του Προέδρου Ομπάμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παροτρύνω τους εταίρους να κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τις κρίσεις στο εξωτερικό ή τον αφοπλισμό, που και αυτό το ανέφερε ο Ομπάμα, ε, στην ομιλία του για την κατάσταση του έθνους ή η ασφάλεια στην αυσιπλοεία, που είναι απειλή στον Ατλαντικό επίσης δεν ήθελα να αφήσω στην άκρη άλλα θέματα, έχετε δίκιο όμως. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα ζήτημα ίσως ε, σημαντικό, αλλά δεν ξέρω το Κογκρέσο πόσο χώρο θα του αφήσει, γιατί είχε executive orders για να προχωρήσει. Εντάξει, θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Το δεύτερο θέμα. Να είμαστε πιο έντονοι ε, στις διατυπώσεις μας προς τη Μέση Ανατολή. Μα σήμερα είναι εκεί ο κύριος Ομπάμα. Το σημείο 27 παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να θέσει ως προτεραιότητα την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε στασιμότητα στη Μέση Ανατολή. Έχει αποτελματωθεί. Παροτρύνει. Τι άλλο να κάνουμε. Ε, ζητάμε να γίνει προτεραιότητα και ένα ε, ε, επαναρχίσουν οι απευθείας διαπραγματεύσεις. Αυτό σας φαίνεται soft. να εξασφαλίσει, λέω, το insurance, σας σας φαίνεται ήπιο αυτό, για τον αφοπλισμό και πάλι στο σημείο 23. Θα προσπαθήσει ο Ομπάμα να κάνει κάποια πράγματα μέχρι και για εσωτερικούς ε, λόγους, ε, γιατί και όχι μόνο με τη Ρωσία για τα πυρηνικά, στο ιστορικό τον είπα υπάρχει λαθρεμπόριο ελαφρού πλεισμού. Στο 23 το λέμε λοιπόν και είμαι βέβαιος ότι με τις τροπολογίες σας ε, θα βελτιώσετε. Το θέμα το θεσμικό. Αυτό το TPC, το θέμα του, του διατλαντικού κοινοβουλευτικού διαλόγου, δεν το βλέπω προς τα μέσο, το βλέπω προς τα έξω. Και εσείς το είπατε και εσείς ε, και ο κύριος Σαλαφράγκα, ο συνάδελφός μου, μιλάτε για τις θεσμικές συνέπειες της συνθήκης ελευθερωση συναλλαγών. Θα υπάρξουν. Και μοιραίο είναι. Θα υπάρχει ένα μεικτό συμβούλιο που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα δίνει κάποια συνέχεια στην εσωτερική, αυτή μεγάλη εσωτερική αγορά. Είναι Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών και θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός θεσμικός παρακολούθησης και διευθέτησης των διαφορών. Υπάρχουν θεσμικές επιπτώσεις, αλλά εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτές. Ε, μιλάω για το πολιτικό διατλαντικό συμβούλιο. Αυτοί δεν ασχολούνται με τα εμπορικά θέματα, θα είναι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών εντό εισαγωγικών, η κυρία Άστον και ο αντικαταστάτη, ο διάδοχός τη, ο κύριο Κέρι και ο διάδοχο του. Η θα δώσει το νέο πλαίσιο, το θεσμικό, αλλά θα υπάρξει συμφωνία ε, εμπορίου και επενδύσεων. Το TPC όμως είναι άλλο πράγμα. Είναι ένα συμβούλιο που θα συντονίζει την εξωτερική πολιτική προς τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, εντάξει, θα υπάρχει και θεσμικές ε, συνέπειες θα έχει και θα δούμε ποιες θα είναι αυτές. Χρειάζεται όμως η δημιουργία μεικτών οργάνων παρακολούθησης, ελέγχου κτλ. Αυτό λέει και ο Σαλαφράγκα. Κύριε Σαλαφράγκα, αγαπητέ συνάδελφοι, χίλια ευχαριστώ, ένα εκατομμύριο ευχαριστώ για τα καλά λόγια και τους επένους ε, που δεν τους αξίζω, είναι μάλλον ε, προϊόν και καρπός της φιλίας μας παρά της δικής μου αξίας. Ε, απάντησα στον κύριο Πιτικόφερ. Πώς βλέπω εγώ τώρα το μέλλον για την τριμερή, αυτή την τριγωνική σύνοδο κορυφής. Προσοχή εδώ. Φέτος δεν το βλέπω για τον εξής προφανή λόγο. Ποιος θα ήταν εκεί, η ΣΕΛΑΚ, ε, η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ στη ΣΕΛΑΚ, προεδρεύει τώρα η Κούβα. Ε, δεν νομίζω να είναι στις προτεραιότητες της ε, κουβανικής κυβέρνησης να έχουμε σε τέτοιο επίπεδο σύνοδο κορυφής τριγωνική με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω μακροπρόθεσμα δεν λέω, δεν αποκλείεται, αλλά είμαι πιο συγκρατημένος. Υπάρχει και μία κόπωση συνόδων κορυφής έτσι και αλλιώς και μετά... Αν δούμε και τι ε, πρεσβεύουν ορισμένοι, δεν είναι στην ημερησία διάταξη της διεθνούς πολιτικής ατζέντα. Ε, το παγκόσμιο διατλαντικό όραμα. Υπάρχουν τα think tank που τα μελετάνε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την ευφία να το πράξει. Η Αγκόλα πουλάει στην Κίνα περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή αυτή η Ατλαντική Αφρική, η Δυτική Αφρική έχει μεγάλο δυναμικό. Και από την άλλη το Μεξικό και άλλοι σήμερα κανένας από αυτούς δεν σκέφτεται με όρους παγκόσμιας ατλαντικής ατζέντα. Σιγά σιγά, πετραδάκι, πετραδάκι. Με αλληλεγγύη, με κάποιες οργανώσεις που λειτουργούν περιφερειακές ως κινητήριες δύναμη και δίνουν την όθηση. Ε, γι' αυτό λέω με την Κεντρική Αμερική ενδεχομένως ε, που αφορά η ασφάλεια και τη ΣΥΠΑ και την Ευρώπη, το θέμα το εμπορικό, το θέμα των ναρκωτικών με την Αφρική και το θέμα το εμπορικό που εμφανίζεται αυτό το τρίγωνο σιγά σιγά. Αλλά εκεί με τις συνόδους κορυφής στρέφονται πιο πολύ προς τον ελληνικό. Εκεί θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε για τον Ατλαντικό χωρίς πολύ μεγάλες προσδοκίες αλλά χωρίς να απεμπολίσουμε και τίποτα και να καλέσουμε τα think tanks, τους ε, ενδιαφερομένους, τις κυβερνήσεις να δραστηριοποιηθούν. Εγώ δεν τρέφω μεγάλες ε, αυταπάτες ούτε προσδοκίες έχω. Ε, σιγά σιγά να μας προβληματίζει να γεννάτε αυτό το ενδιαφέρον για μια συνολική διατλαντική συνεργασία. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2011 ήδη έχει αρχίσει και δίνει σημασία ιδιαίτερη σε αυτό το θέμα. Αυτά. Περιμένω τι τροπολογίε σα και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ. Thank you. Next point. Ευχαριστώ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ενημέρωση από τον Μίλαν Σαμπρνόκ σχετικά με την αποστολή παρακολούθησης των εκλογών στην Αρμενία από τις 16 έως τις 19 Φεβρουαρίου του 2013. Σας υπενθυμίζω ότι στις 18 Φεβρουαρίου έγιναν προεδρικές εκλογές και ο, ο Σέρτ Σαρκοσιάν επανεξελέγει ε, στη χώρα του. Οι διεθνείς παρατηρητές ε, είπαν στην συνέντευξη τύπου ότι οι εκλογές ήταν και παραθέτω γενικά καλά, καλές και ε, ε, σέβονταν τις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Όμως, η αποστολή των παρατηρητών προσέθεσε ότι υπήρξαν κάποια θέματα και ότι, αναφέρω, παρότι η μέρα των εκλογών ήταν ήρεμη και επικράτησε τάξη, στη διαδικασία υπήρξε αν... περιττή αναταραχή λόγω της συμπεριφοράς του Προέδρου. Ο δεύτερος ε, στη σειρά των αποτελεσματών, ο Βάνιο Βανισιάν, ε, έκτοτε συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Στις 2 Μαρτίου η μακροχρόνια αποστολή του ΟΝΤΙΡ εξέδωσε μια έκθεση που είναι πολύ πιο επικριτική και ανέφερε ε, κάποια στοιχεία για το διάστημα μετά τις εκλογές. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Μίλα Ζάπρνοχ που είναι πρόεδρος της ε, Αποστολής Παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να κάνει την αναφορά του σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους του IEOM. Ευχαριστώ. Το, η σωστή προφορά του ονόματό μου είναι Τσάμπνοχ, αλλά δεν πειράζει. Κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε. Σα ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα την τιμή να είμαι πρόεδρο τη αντιπροσωπείας τη αποστολή παρατήρησης των εκλογών, των προεδρικών εκλογών στην Αρμενία στις 18 Φεβρουαρίου. Η αντιπροσωπεία για την παρατήρηση των εκλογών αποτελείται από την ε, κυρία Μπασέσκου, τον κύριο Τσαρνέτς και εμένα τον ίδιο και άλλους δύο συναδέλφους και θέλω να τους ευχαριστήσω για την εξαιρετική μας συνεργασία κατά τη ε, διάρκεια της αποστολής αυτής. Θέλω να επικεντρωθώ εδώ σε δύο σημεία. Οι προεδρικές εκλογές στην Ερμενία πρώτον και η διεθνής συνεργασία στα πλαίσια διεθνών αποστολών παρατήρησης εκλογών. Σε ό,τι αφορά τι πρόσφατε προεδρικέ εκλογέ στην Αρμενία, να θυμίσω ότι οι εκλογέ αυτέ ήταν σαν μία δοκιμή για τον εκδημοκρατισμό της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει πει ρητός στο ψήφισμά του του Απριλίου 2012 κατά τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρμενίας ότι οι ελεύθερες και ανοιχτέ εκλογέ είναι απαραίτητε, πρέπει να είναι διαφανέστερε και να συμφωνούν με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι άκρα σημασία για, την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση-Αρμενία. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ σήμερα έχει να κάνει με την συνεργασία μα στο πλαίσιο των αποστολών παρατήρηση εκλογών. Τέτοιου είδου διεθνεί αποστολέ είναι εχέγγυο ότι η διεθνής κοινότητα θα εκφράζεται με φωνή ενιαία στο πλαίσιο τέτοιου είδους αποστολών. Οι κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ και σε κάποιες περιπτώσεις και του ΝΑΤΟ συμμετέχουν σε τέτοιου είδους, σε τέτοιου είδους διεθνείς αποστολές. Στην Αρμενία η κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ αποφάσισε να μην προσέλθει. Έτσι, εφήρμοσε την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΑΣΕ, από το Δουβλίνο το Δεκέμβριο του 2012, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά του ΑΣΕ με τη χώρα αυτή. Τώρα, ω προ τα ίδια τα γεγονότα και πώ εκτελήθηκαν οι προεδρικέ εκλογέ στην Αρμενία. Συμπεράσματα και συνέχεια που δόθηκε στην όλη διαδικασία. Τα προκαταρτικά συμπεράσματα τη Διεθνού Αποστολή για την Παρατήρηση των Εκλογών είναι ότι ήταν αντικείμενο καλής διαχείρισης η διεξαγωγή των εκλογών και σεβόμενες της θεμελιώδεις ελευθερίες. Το κρατικό, τα κρατικά κανάλια της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου ε, σεβάστηκαν τις βασικές ανάγκες κάλυψης ε, της έκφρασης όλων των υποψηφίων και των ε, τον ισομερή του χρόνου. Βεβαίω, κάποιε στιγμέ υπήρχε μια στρέβλωση μεταξύ κράτου και κυβερνώντο κόμματο, κάτι που αντιφάσκει με το έγγραφο τη Κοπεχάγη που καθορίζει διεθνή πρότυπα για τέτοιου είδου θέματα. Ο ελεύθερο ανταγωνισμό δεν ήταν απολύτω ελεύθερο γιατί τρία από τα μεγαλύτερα κόμματα αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στι εκλογέ, Μετά τη δημοσίευση των επίσημων αποτελεσμάτων που λένε ότι ο πρόεδρο Αρδοσιάν επανεξελέγει ήδη από τον πρώτο γύρο, τότε η αποστολή του ΑΣΕ εξέδωσε την ενδιάμεση έκθεσή της αναφέροντας τις ανησυχίες της για τον στενό συσχετισμό του αριθμού των ψήφων που δόθηκαν στον ε, πρόεδρο και το πώς διοργανώθηκαν τα εκλογικά κέντρα. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο συνταγματικό μάλλον δικαστήριο, με έφεση στις 14 Μαρτίου, αλλά το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και την προσφυγή του και τελικά τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών επικυρώθηκαν. Είναι πολύ σωστό να δίνουμε τέτοια σημασία στη συνέχεια που δίνεται σε τέτοιε διεθνεί αποστολέ παρατηρήσει εκλογών από το Ευρωκοινοβούλιο. Επαναλαμβάνουμε ότι έδειξαν καλή θέληση οι εκλογέ με τις πρόσφατες αυτές προεδρικές εκλογές. Ελπίζουμε όμως να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την ε, υλοποίηση των συστάσεων που έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση της αποστολής με διεξοδικότερη διαδικασία όπου θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί τη κοινωνία. Ενθαρρύνω την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Αντιπροσωπεία για την Κοινοβουλευτική Συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρμενία να ακολουθήσουν τις συστάσεις της έκθεση τη αποστολή μα και να ενημερώσουν αναλόγω τις αρμενικές αρχές. Όπως στην ομιλία μου μετά την διεξαγωγή των εκλογών, είναι καθοριστική σημασία οι αρμενικές αρχές να δώσουν περαιτέρω αποτελέσματα για την πρόθεση του εκδημοκρατισμού και των πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητε για την ε, σύναψη Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Αρμενία. Κάτι που θα καθορίζει και το μέλλον των επόμενων εκλογικών διαδικασιών. Πρόεδρε, να κλείσω λέγοντά σα ότι ανησυχώ ιδιαίτερω για τη θέση τη κοινοβουλευτική συνέλευση του ΟΑΣΕ. Βρίσκω ότι είναι ατυχής και επιζήμια από πολλές απόψεις η θέση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης σε επίπεδο ΟΑΣΕ πλήττει το δυναμικό, τη δυνατότητα της διεθνούς κοινότητας να εκφράζεται με ενιαία φωνή. δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοια διαφωνία μεταξύ των ε, συμμετεχόντων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή του ΑΣΕ. Θα πρέπει η Ρωσία, το Καζακστάν, η Λευκορωσία, η Αρμενία, το Κυργιζιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν, οι, συμμετέχοντες, οι συμμετέχουσες αυτές τις χώρες, να πάψουν να αποδυναμώνουν το ΟΝΤΙΡ. Και την δυνατότητα παρατήρησης ε, εκλογών εδώ, έχουμε επανειλημμένως απευθυνθεί στην ΟΑΣΕ ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω το τμήμα αυτό του ΑΣΕ, το δύρ και να μπορέσουν ε, οι αρμόδιοι φορείς του ΑΣΕ να παρατηρούν αποτελεσματικά τις εκλογές. Τα συμπεράσματα του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης θέτουν σε κίνδυνο την ε, εργασία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς το Ευρωκοινοβούλιο ανέκαθεν υπερασπιζόταν τέτοια θύματα μεγάλη σημασία και για τον εκδημοκρατισμό και για το κράτος δικαίου. Η ομάδα συντονισμού και παρατηρήση εκλογών, όπου συμπροεδρεύει ο κύριος Μπροκ, συναντήθηκε στις 26, θα συναντηθεί μάλλον στις 26 Μαρτίου, για να ανταλλάξουμε ε, στοιχεία για τα θέματα αυτά. Θα παραστεί και ο κύριος Μακμίλαν Σκοτ και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα βρει τρόπους να επηρεάσει ώστε να διορθωθεί αυτή η ατυχής κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Δεν υπάρχει κάποιος ε, συνάδελφος να δέχεται το λόγο. Οπότε, το επόμενο σημείο είναι... Σας ευχαριστώ και πάλι για την ε, παρουσίαση αυτή ενημέρωση από τον κύριο Λίζε και τον κύριο Πέτερλε για την αποστολή παρατήρησης εκλογών στην Κένια στις 2 6 Μαρτίου 2013. Χαίρομαι πολύ που και ο κύριος Λίζε που ηγήθηκε της ε, μήνυ αυτής αποστολής καθώς και ο κύριος Πέτερλε βρίσκονται εδώ. Οι εκλογές διεξήχθηκαν την Δευτέρα 4 Μαρτίου και ως τώρα τα... η διεξαγωγή τους κρίθηκε ειρηνική και ήρεμη. Όχι όπως τις προηγούμενες εκλογές το 2007 με τα βία γεγονότα. Βεβαίως ήταν μικρή η διαφορά για την νίκη του κυρίου Κενιάτα και του συνασπισμού του, η οποία δέχτηκε βέβαια νομική προσφυγή εναντίον της. από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχουν ε, κατηγορηθεί ανοιχτά ο κύριος Κενιάτα και άλλα μέλη του συνασπισμού του. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για την επίσκεψη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε ότι το γεγονός ότι συναντιόμαστε εδώ με τον κύριο Πίτερλε επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό που ήθελα να πω, ότι η συνεργασία δηλαδή σε τέτοιου είδους ε, αποστολές παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αποστολής που ήταν κεφαλής ο κύριος Πέτερλε και η συνεργασία με τη δική μας αντιπροσωπεία που βρέθηκε εκεί μόνο για δύο μέρες ήταν εξαιρετική. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Πέτερλε επειδή θεωρώ ότι καταφέραμε να συνεργαστούμε πολύ καλά. Μας φρόντισε. Όπως είπα, η δική μας αποστολή ήταν πολύ σύντομη διάρκεια. Μπορούμε λοιπόν να αναφερθούμε μόνο συγκεκριμένα στην τελευταία μέρα της προεκλογικής εκστρατείας και βεβαίως να αξιολογήσουμε μόνο κάποιες από τις βασικές συναντήσεις που είχαμε με, την, με τις υπηρεσίες που ήταν υπεύθυνε για τις εκλογές και κάποιους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Τέτοιου είδους συναντήσεις είχα. είχαμε φυσικά με το διπλωματικό Σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους μόνο δύο φορές. Η δική μας αντιπροσωπεία αποτελείται από 7 μέλη. Εκπροσωπούσαμε 6 χώρες, 7 διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Αισθάνομαι λοιπόν ότι παρά το ότι η αποστολή ήταν σύντομη και η ομάδα μας ήταν μικρή, είχαμε ευρεία εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών του ομάδων. Όπως σας είπα, εισαγωγικά, η αποστολή ήταν σύντομης διάρκειας, γιατί μείναμε εκεί για λίγο μόνο διάστημα. Μας φρόντισε ο κύριος Πέιτερλε, μας ε, παρήχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ευθύς εξ αρχής και έγιναν διάφορες ε, συναντήσεις με διαφόρους εκπροσώπους της Κένιας. Πρέσβεις, σχεδόν όλους τους πρέσβεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνται εκεί με πρέσβεις νομίζω ότι συνολικά ήταν 17 αρκετοί και όλοι παραβρέθηκαν σε συνεδρίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα οι συνεδρίες, παρότι μερικές φορές διαπιστώσαμε ότι οι πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ε, διστάμενες απόψεις επί κάποιων θεμάτων. Όπως σας είπα λοιπόν, καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους από τους υποψηφίους ε, και του Προέδρου. Δεν μπορέσαμε όμως να ε, συναντηθούμε, επειδή ήταν σύντομη η διάρκεια της παραμονής μας εκεί, δεν μπορέσαμε να ε, συναντηθούμε με τους βασικούς υποψηφίους. Επ' αυτού θα μας ενημερώσει καλύτερα ο κύριος Πέτρελε. Όπως είπα, συναντηθήκαμε με τους υπεύθυνους για την οργάνωση των εκλογών, όπως και με εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων. Την ημέρα τώρα των εκλογών, η ομάδα μας χωρίστηκε σε τρία μέρη και παρακολουθήσαμε τις εκλογές στην πρωτεύουσα, στο Ναρόμπι, όπως επίσης και στην, στο Ναϊβάσο που είναι στο βόρεια του Ναϊρόμπι, σε μια ε, περιοχή της Υπέθρου και από τις παρατηρήσεις μας κατά την ημέρα των εκλογών και όλα αυτά περιγράφονται στην έκθεση γνωμοδότησης που σας έχουμε ήδη συνάδουν με τις ε, παρατηρήσεις του κυρίου Πέτρελε. Θα αναφερθώ λοιπόν σε αυτό τα οποία είδαμε εμείς με τα μάτια μας την ημέρα των εκλογών. Στα δύο αυτά μέρη που πήγαμε για να παρακολουθήσουμε τις εκλογές, οι εκλογές ε, ήταν οργανωμένες καλά και όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας μας επεσήμαναν τον μεγάλο επαγγελματισμό και την ε, προετοιμασία των μελών της ε, Επιτροπής Οργάνωσης των Εκλογών. Τα μέλη ε, των φορευτικών επιτροπών στα εκλογικά κέντρα ήταν καλά προετοιμασμένα, δεν, μας υποδέχτηκαν καλά, δεν υπήρξε παραμικρή επιφύλαξη ούτε από δική μας πλευράς, ούτε και από τους άλλους πολλούς παρατηρητές, ντόπιου ή διεθνείς που ε, παρακολουθούσαν τις ίδιες εκλογές. Όπως και εσείς κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε στον προηγούμενο γύρο εκλογών τότε την ημέρα των εκλογών είχαν ε, συμβεί μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Όταν όμως εμείς βρισκόμασταν εκεί, μόνο ένα ατυχές γεγονός συνέβη στη Μομπάσα. Δυστυχώς υπήρξαν και θύματα απώλειες ζωής, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ανθρώπων που δούλευαν στα στους εκλογικά κέντρα αστυνομικών και μελών του Ρυθρού Σταυρού. Η κατάσταση στη Μομπάσα όμως δεν είχε καμία σχέση με τις εκλογές. Αυτό ήταν ένα επεισόδιο που προκλήθηκε από τη δράση μιας ομάδας αποσχιστικής που θέλει να ε, αποσχιστεί ένα ολόκληρο μέρος της Κένιας από τη χώρα. Αποφάσισαν την ημέρα αυτή των εκλογών να εκφράσουν τα αιτήματά τους. Όπως σας είπα ήταν μια τραγική, ένα τραγικό επεισόδιο επεισόδιο τοπικής όμως εμβέλεια που δεν διαχύθηκε στην υπόλοιπη χώρα και υπήρξαν δεν υπήρξαν άλλου τέτοιου είδους καταστάσεις στον Ναϊρόμπι ή οπουδήποτε αλλού. Όπου ήμασταν εμείς η κατάσταση ήταν ειρηνική. Προς μεγάλη προς έκπληξη κάποιων από εμά και των Κενιατών δώσαμε την άποψή μας και επισημάναμε ότι υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές ενδεχομένως εσείς θα έχετε εμπειρία από άλλες χώρες και άλλες υποστολές παρατηρητών. Φανταστείτε όμως τις ουρές στην Πολωνία. Εδώ τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έγιναν ουρές ε, στην Κένια από τις 3 ή 4 το πρωί και τα πολιτικά κόμματα προφανώς έκαναν έκκληση να υπάρξει συμμετοχή στις εκλογές. Ε, οι άνθρωποι πήγαν στα εκλογικά κέντρα, περίμεναν ήρεμα, ήσυχα, χρειάστηκε να περιμένουν επί ώρες και σε κάποιες ουρές υπήρξαν μέχρι και χίλια άτομα που περίμεναν ε, για να ψηφίσουν. Όμως, παρά τα μικρά αυτά προβληματάκια, οι εκλογές αυτές καθεαυτές πήγαν καλά και ε, ήρεμα. Αυτά τα οποία ε, είδαμε και το παρατήρησαν και άλλες αντιπροσωπείες παρατηρητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τοπικοί παρατηρητές ε, ήταν ότι ήταν ε, ένα φιάσκο το θέμα της, του ενός πολύ προηγουμένου ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές για τις αναγνώριση. Αυτό δεν λειτουργήσε πολύ καλά και που είχε εγκατασταθεί σε κάποιες ε, περιοχές ε, λειτουργήσε μόνο για λίγες ώρες, αλλού δεν λειτουργούσαν οι μπαταρίες και δεν υπήρχε ηλεκτρικό. Ε, αυτές ήταν μικρές δυσκολίες, αν θέλετε, στην τεχνικής φύσεως. Στην ε, συνέντευξη τύπου που ακολούθησε όμως είπα ότι σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει τέτοιο ηλεκτρονικό σύστημα τόσο προηγουμένο. Πάση περιπτώσει. Τώρα, οι, οι επιτροπές, ε, τα εκλογικά τμήματα, όλα λειτουργήσαν καλά και γρήγορα και επέστρεψαν στο πιο παραδοσιακό σύστημα αναγνώρισης των ψηφοφόρων, κοίταζαν τα ονόματα, τα διέγραφαν δεν χρειάστηκε να πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα από αυτούς που πήγαιναν να ψηφίσουν, αλλά εν γέννη και συνολικά όλα λειτουργήσαν. Ένα σημαντικό ζήτημα που θέλω να υπογραμμίσω είναι οι προεκλογικές συναντήσεις που κάναμε. Ο κύριος Κενιάτα ήταν υποψήφιος Θελήσαμε να τον συναντήσουμε, αλλά δυστυχώς απορρίφθηκε το αίτημά μας, αρνήθηκε να συναντηθεί με την προσωπία μας. Υπάρχει ένας πολιτι... μια πολιτική... ένας πολιτικός χώρος γύρω από τον κύριο Οντίνγκη. Ε, από αυτούς καταφέραμε να συναντηθούμε με ένα σημαίνον στέλεχος της, τον επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας, ο οποίος υπογράμμισε στις επαφές μας ότι αυτό το πολιτικό στρατόπεδο θα σεβόταν το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως επίσης και οποιαδήποτε απόφαση των δικαστηρίων. Γιατί θα διαβάσατε και στον τύπο ότι αυτό έχει αναφερθεί εκτεταμένα σήμερα βλέπουμε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η διαδικασία αυτή. Η Επιτροπή Κλογών, όμως ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Ε, έχει ένα ποσοστό 0,4%. Ε, θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι από τα εκατομμύρια των ψήφων το αποτέλεσμα αυτό προσωπεί μόνο κάποιες χιλιάδες και έχει αμφισβητηθεί. Τώρα λοιπόν τελικά περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι η απόφαση θα βγει σε περίπου μία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Πέτερλε έχει κάποια ε, πιο πρόσφατη ενημέρωση από ότι εμείς. Εμείς αυτά γνωρίζουμε. Εξ όσων γνωρίζω λοιπόν, εισαγωγικά αυτά έχω να πω και βεβαίω αν έχετε ερωτήσεις με τα χαρά θα σας απαντήσω. Ο κύριος Πέτρος όμως έχει ε, περισσότερη λεπτομερή ενημέρωση γιατί ήταν επικεφαλής μιας επιτροπής που και μεγαλύτερο διάστημα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήμουν και εγώ στην αποστολή αυτή όπου ηγήθηκε ο κύριος Λίζε, ο οποίος ήταν όχι μόνο πολύ αποτελεσματικός στη διοργάνωση μιας ομάδας των βουλευτών, αλλά ήταν και πολύ καλός, είχε πολύ καλή μνήμη. Η έκθεση που υπέβαλε είναι ιδιαίτερα δεξοδική, αλλά θέλω να προσθέσω τα εξή. Όπως είπατε, πριν από πέντε χρόνια οι εκλογές ήταν τραγικά διαφορετικές Περίπου 200.000 έχασαν τη ζωή τους, 5.000 ε, εκτοπίστηκαν και πολλοί είναι αυτοί που βρέθηκαν ε, εκτός των αισθειών τους. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάρτισε τέτοιες εκθέσεις που σημείωνε τι εξελίξει, ιδίω όταν άλλαξε ο εκλογικό νόμο και όταν έγιναν συνταγματικέ μεταρρυθμίσει. Η Κένια, λοιπόν, από νομική πλευρά ήταν σαφώ ετοιμότερη για την σωστή διεξαγωγή των εκλογών. Ο εκλογικό νόμο είχε αλλάξει, το Σύνταγμα είχε μεταρρυθμιστεί, υπήρχε ανεξάρτητη εφορευτική επιτροπή ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία η ανεξαρτησία του επίση είχε μεταρρυθμιστεί το δικαστικό σύστημα εντωμεταξύ, το δικαστικό σώμα και στην ουσία υπήρχαν έξι εκλογέ ταυτόχρονα Προεδρικέ, περιφερειακέ, τοπικέ. Όλε ταυτόχρονα. Αυτό ήταν μια σημαντική πρόκληση και για του ε, ψηφοφόρους, αλλά και για τις εφορευτικές επιτροπές. Πάντως, τα πάντα έγιναν με, άκρα, με μεγάλο επαγγελματισμό με κάποια μικρά τεχνικά προβλήματα, όμως για τόσο βαρύ πρόγραμμα εκλογών τα πάντα πήγαν αρκετά καλά. Τα αποτελέσματα τα ακούσατε, όμως ήταν πολύ μικρή διαφορά για τον νικητή, 0,7%. Είναι στην πραγματικότητα εκατοντάδε χιλιάδε οι ψήφοι που χωρίζουν τον κύριο Κενιάτα από τον κύριο Ουδίνγκα. Ο συνασπισμό του κύριου Ουδίνγκα έχει προσφύγει ήδη από το Σάββατο, άρα για μα δεν είναι τελεσίδικη η έκβαση. Σε δύο εβδομάδε θα εξεταστεί η προσφυγή και το δικαστήριο θα πρέπει να εκδώσει απόφαση. Όμως, η πλευρά ε, που προσέφυγε θέλει να ακυρωθούν ε, οι εκλογές συνολικά. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου βλέπουμε με ικανοποίηση ότι παρόλα αυτά τα πράγματα προχωρούν ειρηνικά. Όλοι οι βασικοί συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία έχουν καλέσει τους ε, υποστηρικτές τους να εκφράζονται και να διαδηλώνουν εάν χρειαστεί, ειρηνικά. Πολλοί είναι εκείνοι που προέβλεπαν ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν αρκετά διαφορετικά. Κάποιοι, μάλιστα, έφυγαν τρέχοντας από τον Αερόμπι και την Κένια, φοβούμενοι ότι μπορεί να συμβεί ποιος ξέρει τι. Όμως, η Κένια έδειξε ότι έχει οριμάσει. Ελπίζουμε ότι αυτό θα εξακολουθήσει και μετά την έκδοση τη απόφαση του δικαστηρίου. Να πω ότι η αποστολή μας δεν είχε καθόλου ρομαντικό χαρακτήρα. Είχαμε 65 συμμετέχοντες, όμως κάποιοι αφισβήτησαν την αντικειμενικότητά μας και την αμεροληψία μας. Συχνά χρειάστηκε να συστηθούμε, να εξηγήσουμε ποια ακριβώ είναι η αρμοδιότητά μα, ποια η εντολή που έχουμε αναλάβει, αλλά με την συνεργασία όλων καταφέραμε να πείσουμε τους πάντες ότι είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί. Τέθηκε όμως και στη συνέντευξη τύπου ένα άλλο θέμα που ανέκυπτε επανειλημμένος και αυτό ήταν τι πιστεύουμε για το γεγονός ότι δύο από του υποψηφίου ε, στι εκλογέ κλήθηκαν ενώπιον του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Βέβαια, δεν είχαμε καμιά πολιτική εντολή να πάρουμε θέση και να εκφράσουμε πολιτικέ προτιμήσει. Όμω, εάν το ζήτημα αυτό ε, αποτελέσει θέμα στην όλη πολιτική διαδικασία, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντω, ε, κατά τη διάρκεια τη εκλογική διαδικασία, δεν θέλαμε να παρέμβουμε καθόλου και να τοποθετηθούμε. Τα πράγματα λοιπόν πήγαν περίπου όπως σας είπα και όπως είπε ο κύριο Λίζεκ. Υπάρχουν κάτι μέλη με διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα, απόψεις που όμως έχουν εκφραστεί και ούτω ή άλλω ήταν εκλογέ που προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν τόσο πολλοί παρατηρητέ που συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή. Η Αφρικανική Ένωση πραγματικά έκανε μια τολμηρή προσπάθεια, μια αξιέπαινη προσπάθεια για να συντονίσει την αποστολή των συντονιστών, οι οποίοι πραγματικά συνεργάστηκαν αρμονικά και συνεισέφεραν στο να μπορέσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Γι' αυτό είχαμε καλά αποτελέσματα. Συναντήσαμε πολλούς υποψηφίους, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους του συναπλισμού του κυρίου Κενιάτα, και τον κύριο Ρούτο συναντήσαμε, τον ε, υπαριθμών 2 στο συνασπισμό. Και μάλιστα ακολουθήσαμε τη διαδικασία με μεγάλη προσήλωση στους τύπους. Συνομιλήσαμε με όλους τους υποψηφίους με τον ίδιο τρόπο. Προκειμένου να είμαστε βέβαιοι για το πόρισμα ότι οι εκλογές είναι αδιάβλητες και ελεύθερες. Βεβαίω, απόφαση δικαστηρίου ακόμη δεν έχει εκδοθεί και πριν ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο τη διαδικασία, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε οριστικά. Αυτέ είναι οι δικέ μου παρατηρήσει. Υπάρχουν και άλλε ενδιαφέρουσε λεπτομέρειε. Γιατί πολλοί είναι αυτοί που μας αμφισβήτησαν, αλλά σε γενικές γραμμές καλοδεχούμενοι αισθανθήκαμε. Απλώς Κάποιοι θέλανε να παρέμβουμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό δεν ήταν ε, μέρος της εντολής μας. Ευγενικά τους παραπέμπαμε στους αρμοδίους. Και ολοκληρώνοντας την ε, δική μου παρέμβαση, να πω ότι διδάχτηκα πολλά από την Κένια. Έμαθα πολλά για τη χώρα. Μπορεί να είναι ένας αξιόλογος εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και μπορούμε να δούμε τι μπορεί να σημαίνουν εκλογέ εκλογές και σε τοπικό και σε διεθνέ επίπεδο. Παράλληλα, οι γείτονε χώρες είχαν καταστήσει σαφή και τη δική τους στάση. Θέλαν να διεξαχθούν με ειρηνικό τρόπο εκλογές. Αυτά από μένα και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Υπάρχει κανείς που να θέλει το λόγο. Ο κύριος Γκερέρο. Yeah, the floor. Sí. Ναι, ευχαριστώ. Ναι, κοιτάξτε, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι αισθάνομαι ότι και ε, τα όσα είπε ο κύριος Λίσα και τα όσα είπε ο κύριος Πέτερλε με αντιπροσωπεύουν πλήρως και στις δύο περιπτώσεις πραγματικά με τρόπο σαφή όσο και αντικειμενικό ε, αντανακλούν τα όσα πράξαμε εμείς στην Κένια. Και το αποτέλεσμα θα δούμε ποιο θα είναι μόλις εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου και ελπίζουμε να είναι ειρηνική έκβαση αυτού που ήταν σύραξη πραγματικά το παρελθόν. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι μετά από αυτή τη μακρά ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και για την προσοχή σας και κυρίως το πέρα της συνεδρία